του Γενικού ε, Δικαστηρίου μου είχε ζητήσει διοικητικά στοιχεία ε, και του τα χρωστάω γιατί του τα έχω υποσχεθεί. Κάνω μια, πα, μια παρένθεση για το Brexit. Δεν ξέρουμε φυσικά ποιες θα είναι οι συνέπειες ε, του Brexit στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι ιδιαίτερα πολιτικό και λεπτό το ζήτημα. Ξέρετε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία τα πιο πολεμικά στην ε, συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν θα υπάρχουν ε, πλέον προδικαστικά ερωτήματα που θα στέλνονται από τους Βρετανούς δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν υπάρχουν πολλά, θα, θα είναι λιγότερα. Δεν ε, θα υπάρχει ουσιαστικά προσφυγή λόγω παραβαση ε, που ε, θα καταθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν ε, θα έχουμε ουσιαστικά μειωμενε υποθέσεις στα αγγλικά. Τώρα αν θα έχουμε και λιγοτερε υποθεσει στο δικαστήριο, εγώ πιστεύω πω όχι, γιατί πιστεύω ότι θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει μια διαφορά που θα ε, εμφανιστεί και θα σχετίζονται με τον Brexit, δηλαδή πολίτες ε, που θα ζουν στην Ισπανία ή σε κάποια άλλη χώρα και θα απευθυνθούν στον Ισπανό δικαστή για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και αυτό θα καταλήξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγώ υποθέτω ότι υπάρχουν ε, περισσότερες υποθέσεις αλλά λιγότερες στην αγγλική γλώσσα. Θα εξετάσουμε λοιπόν περισσότερο το στοιχείο αυτό για το θέμα της ενδεχόμενης ε, αλλαγής ε, της γλώσσας των διασκέψεων, όμως ε, το δικαστήριο, αν το επιθυμεί, θα μπορέσει, να θα μπορέσει να αποφασίσει σε ποια γλώσσα θα εργαστούν οι δικαστές μεταξύ τους, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και ήδη μίλησα για το σύστημα πληροφορικής, τώρα να πάμε στα άλλα ζητήματα έχω απομακρυνθεί τόσο πολύ που μπορεί να τα ξεχάσω. Λοιπόν, ε, θα φτάσω και στο θέμα της παρουσίας των γυναικών. Ε, ευχαριστώ που μου δώσατε και τα στοιχεία. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουμε πέντε γυναίκες δικαστές ε, και δύο γενικές εισαγγελίες μεταξύ των 39. τώρα, στην μεταρρύθμιση Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε να αυξηθούν οι γυναίκες δικαστές στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν εξαρτάται ε, μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν εξαρτάται καθόλου από το δικαστήριο. Οι άνθρωποι που προτείνονται, προτείνονται από τα κράτη-μέλη. Εμείς ε, ευχαρίστω να έχουμε όλο ένα και περισσότερε γυναίκε. Ε, αν ισχύσει, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τα δυσιομενικά για τον προπολογισμό. Να πάω στον κύριο Μαρίνιο Πίντο. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία διαθέσιμα. Μπορούμε να τα προσθέσουμε βέβαια. Έχετε όμω διάφορα στοιχεία στη διάθεσή σα. Θα ήθελα, θα ήθελα αναλυτική πληροφόρηση ο κύριο Μαρίνιο Πίντο. Να υπενθυμίσω όμως το εξή. Ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί το 4% του προπολογισμού των διοικητικών δαπανών της Ένωσης. Είναι το 4%. Αυτός ο αριθμός ε, μένει σταθερός εδώ και χρόνια. Στην πραγματικότητα μάλλον έχει μειωθεί. Το 2010 είμαστε στο 4,13 ενώ τώρα είμαστε στο 4% μετά τη μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ο προπολογισμό τη δικαιοσύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να το πω για να σα δώσω κάποιε αποχράσει. Επίσης, η μεταρρύθμιση που κράτησε τόσα χρόνια από το Μάρτιο του 2011 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ε, το δικαστήριο προσπαθούσε να ανταπεξέλθει ε, σε όλο αυτό τον όγκο εργασίας με μη επαρκή αριθμό δικαστών και ε, για το έτος 2017 είχαμε 3,4 αύξηση του προπολογισμού, για το 2018 θα έχουμε 3,32. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τίμημα για τη δικαιοσύνη, υπάρχει ένα τίμημα, αλλά είναι λογικό το τίμημα σχετικά. Μιλήσαμε για τους εισηγητές. Με συγχωρείτε. Ε, εμείς είχαμε σχεδιάσει μέχρι τις 4 την, πρώτη, ε, την συνεδρίαση αυτή, την κοινή αυτή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Άρα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ και απλώς ε, σας παρακαλώ να το σημειώσετε. Μπορώ να σταματήσω και εδώ αν θέλετε κύριε Πρόεδρε. Απαντάω ο κ. Σκομπάρ. Ε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αλλά άλλα μέλη έχουν λάβει απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν. Σεις κυρία Χάουταλα επιθυμείτε να λάβετε το λόγο. Άκουσα ότι είπατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει περισσότερους δικαστές. Από όσο ξέρω, κάναμε μια διοργανική δήλωση. Άρα όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απογοητευθήκαμε ιδιαίτερα όταν είδαμε τις πρώτες, τους πρώτους διορισμούς μετά από αυτό που θεωρώ ότι δεν ήταν ε, έντιμο παιχνίδι. η πρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ για τι εξηγήσει σα. Αν δεν ήσασταν σημαντικοί, δεν θα καθόμασταν εμεί εδώ σήμερα μαζί σα. Και εμεί τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού συζητήσαμε, α το πω έτσι διπλωματικά, συζητήσαμε επί μια τριετία για το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω και ορισμένε ερωτήσει, αλλά θα σα τι στείλω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρακαλώ να μου απαντήσετε γραπτώ. Αλλά σα ανακοινώνω από τώρα ότι στα πλαίσια της ετήσια συζήτησης για την απαλλαγή του προϋπολογισμού θα επανέλθουμε σε ερωτήσεις αυτές. Δεν μπορούμε να φανταστούμε καν να αντικαταστήσουμε τη γαλλική γλώσσα από την αγγλική και την λέω, τα λέω αυτά στα γαλλικά διότι νομίζω ότι μιλώ καλά γαλλικά. Δεν θα πρέπει να μεταφράζονται τα κείμενα από τα αγγλικά στα γαλλικά και μετά να επαναμεταφράζονται στα αγγλικά. Πρέπει να επιτρέψουμε να λειτουργούν διάφορες γλώσσες, τουλάχιστον αυτές οι δυο, γιατί δεν εξυπηρετεί η μετάφραση για να ε, δικαιωθεί μόνο αυτή η απόφαση των δικαστών του 1952. Αν και έστω και αν υπάρχει σε ένα κείμενο του 1952. Ε, θα ασχοληθούμε με αυτό και ε, ευχαρίστως θα σας ξανασυναντήσουμε. Πρόεδρος, δυστυχώς και εάν το ελεγκτικό συνέδριο δεν θέλει να πει κάτι το απολύτως αναγκαίο για να απαντήσει στα όσα είπε το δικαστήριο. Όχι λοιπόν, καλώς. Θα σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ όλους και τις δύο αντιπροσωπείες από το ελεγκτικό συνέδριο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έλευση σας εδώ και για τις διευκρινήσεις που δώσατε. Ευχαριστώ. Κλείνει ε, ε, λίγη η κοινή συνεδρίαση. Προτείνω να συνεχίσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τη μερσία διάταξη. Ένα θέμα παραμένει για σήμερα το απόγευμα η προληπτική αναδιάθρωση, δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναδιάθρωσης, αφαιρεγκαιότητα και απαλλαγή. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, χαίρομαι που τα καταφέρνουμε σήμερα το απόγευμα να μιλήσουμε για αυτή τη σημαντική ε, πρόταση οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαρίστω δε να τα συζητήσω με του συναδέλφου μου. Περί τίνο πρόκειται. Διαβάσατε τον τίτλο. Πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για ε, μέτρα προληπτικής αναδιάρθρωσης, την δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης. Είναι βέβαια κάπως βαρύς ο τίτλος, αλλά ε, με λίγα λόγια πρόκειται περί του εξής. Με το ρυθμιστικό πλαίσιο στοχεύεται να δοθεί στα χέρια των εταιριών ένα εργαλείο, ένας μηχανισμός που να επιτρέπει να απο, να, να τους επιτρέπει δηλαδή να αποφεύγουν την πτώχευση. Άρα, να έχουν στη διαθέσή τους ένα αριθμό μέτρων ώστε να μπορούν να αδιαρθρώνονται, να αναδιαρθρώνονται και να έχουν την ευκαιρία να συνεχίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με επιτυχία. Αυτό θα ωφελήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, θα ωφελήσει τους εργαζομένους, καθώς και τους εργοδότες βεβαίως, βεβαίως για να διατηρηθούν και θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη ότι ε, υπάρχουν άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι ευκολότερο να απαλλαγεί κανείς από χρέη και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Αν λοιπόν είναι δυνατόν σε μια νεοφυή επιχείρηση για παράδειγμα, η οποία ενδεχομένως να μην ε, τα καταφέρει, να μην ε, βαρύνεται ο επιχειρηματίας για όλη τη ζωή με τα χρέη που έκανε από την ε, ατυχή αυτή προσπάθεια να του δοθεί έστω και σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας, μια δεύτερη ευκαιρία να αναλάβει ξανά επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεύτερη ε, παρατήρηση. Έχω διεξαγάγει πολυαριθμότατες συζήτησεις, διότι χρειάστηκε να πολυδοσκοπήσω πάρα πολλές ομάδες ε, συμφερόντων. Βεβαίως είναι τα συμφέροντα αφενός της επιχειρήσεως, αφετέρου των εργαζομένων, των προμηθευτών, απέναντι στους οποίους υπάρχουν δεσμεύσεις είναι οι ομάδες των πελατών, υπάρχουν οι πιστωτές. Υπάρχει λοιπόν ένας μεγάλος αριθμός συμφερόντων που όλα αυτά οφείλουν να ληφθούν υπόψη. Στην βάση των πολλών αυτών συζητήσεων που έκανα και εγώ και οι συνεργάτες μου, μπόρεσα να περιλάβω και κάποιες τροπολογίες στην έκθεσή μου για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι ένα έντιμο συμβασμό αυτό που προτείνω. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τι προτάσει των συναδέλφων μου, διότι βεβαίω αυτό που χρειάζεται στην πραγματικότητα είναι σωστή εξιστα... ε, ε αντιστάθμιση, ε, ε, εξισορρόπηση των ε, διαφορετικών συμφερόντων. Όπως είπα, υπάρχουν τροπολογίες. Έχω θέσει κατ' επανάληψη την ερώτηση πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον έντιμο έμπορο, τον έντιμο επιχειρηματία. Πώς θα μπορέσουμε να τον διακρίνουμε από τον επιχειρηματία εκείνο ο οποίος έχει τόσες φορές ξαναπέσει στα κόκκινα νούμερα, στο παθητικό δηλαδή, που δεν υπάρχει πλέον ε, καμία πιθανότητα να μπορέσει να ανακάμψει. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια διαδικασία που θα είναι καθαρό, ότι πρόκειται για έναν έντιμο επιχειρηματία ο οποίος έχει μια πραγματική προοπτική εξυγίανση της επιχείρησής του ή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και να αποφύγουμε να, πέσουν ε, να πέσουμε σε επιχειρήσεις οι οποίες θα εκμεταλλευτούν τους κανόνες αυτούς για να ε, προχωρήσουν σε παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι σκέψεις με καθοδηγούσαν. Μετά από αυτά τα προκατακριτικά λόγια θέλω να πω ότι μέσω των τροπολογιών μου θέλω να τονίσω ότι θεωρώ σκόπιμο και για διαδικασίες αναδιαθρώσεως αυτές να εποπτεύονται, να επιτηρούνται αν θέλετε από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και όλα εντός των προθεσμιών και θεωρώ ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν συμφωνήσει τουλάχιστον η πλειοψηφία των δανειστών ή των πιστωτών ε, για την διαδικασία αναδιάθρωσης. Και όταν μιλώ για την πλειοψηφία των ε, ε, δανειστών της επιχείρησης, για μένα είναι αναγκαίο σε αυτούς να συγκαταλέγονται και οι εργαζόμενοι. Και βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα της επιχείρησης και να συμμετέχουν και αυτοί. Κάτι που δεν μπόρεσα να επιλύσω μέσα στο σχέδιο της εκθεσής μου, που ελπίζω όμως να προκύψουν κάποιες λύσεις μέσα από τον συζητήσεων με τους συναδέλφους, είναι τι θα κάνουμε με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις με βιοτεχνίες, με τεχνίτες, με πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, διότι στις ακροάσεις και συζητήσεις που διεξήχθησαν, ακούσαμε συχνά και ξεχνά ότι χρειάζονται ειδικέ ρυθμίσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είμαι απολύτω ανοιχτή σε προτάσει. Αλλά δεν έχω προβλέψει ειδικέ ρυθμίσει για πολύ μικρέ επιχειρήσει. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθούν τέτοιε μέσω των τροπολογιών. Ίσως μπορέσουν να προκύψουν κάποιες αρχές λύσεων. Έρχομαι στην έκθεση. Θα διεξέλθω τα διάφορα σημεία, τις διάφορες ε, παραγράφους. Έχω στην παράγραφο 3 την έγκαιρη προειδοποίηση. Εδώ νομίζω είναι κάπως αόριστη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό προσπαθώ εγώ εδώ να διευκρινίσω πώς θα διαμορφωθεί πιο συγκεκριμένα ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και διατυπώνω και μία εντολή προς εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την πορεία της επιχείρησης να αναπτύξουν κάποιους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. Δηλαδή όταν η πλευρά των πιστωτών βλέπει ότι αρχίζει και ε, σιωρεύει οφειλές η επιχείρηση, θα πρέπει να κινητοποιηθεί και προς το ίδιο συμφέρον η ομάδα των πιστωτών για να ε, βάλει μπροστά τους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης. Άρθρο 4. Αναφέρεται στην διαθεσιμότητα προληπτικών μέτρων αναδιάρθρωσης. Εδώ βλέπω να λείπει στην πρόταση της Κομισιόν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να ληφθεί μια απόφαση, δηλαδή πότε αρχίζει να κινείται ο μηχανισμός. Είναι αόριστη διατύπωση εδώ. Εγώ πήρα αυτό το likelihood of insolvency, πιθανότητα δηλαδή ε, να το διευκρινίσω κάπως περισσότερο, να το ορίσω καθαρότερα. Ε, αν έχετε ε, προτάσεις, πολύ ευχαρίστω να τις ακούσω. Άρθρο 5, ιδιοδιαχείριση οφειλετών. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσουν οι στον τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων όσο αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει να προβλέπεται ωστόσο διορισμός συνδίκου για την διαχείριση. Από τις πολλές συνομιλίες που έκανα έμαθα, αλλά δεν το έχω ε, επαληθεύσει γιατί εμπειρικά μου είπαν ότι υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, insolvency practitioners δηλαδή, μου είπαν ότι 80% των περιπτώσεων αφαιρεγγιότητας, που καταλήγουν δηλαδή επιχειρήσει αφαιρεγγιότητα, οφείλονται σε λάθη της διαχείρισης. Εάν αυτό συμβαίνει, μόνο η διαχείριση, το, το management δηλαδή, είναι σε θέση πράγματι μόνο του να κάνει την αναδιάρθρωση ή υπάρχει πραγματικά ρόλος να του προσφέρει συνδρομή κάποιος, όχι απαραίτητα, μάλλον καθόλου διορισμένος από το δικαστήριο, αλλά κάποιος ο οποίος έχει γνώση των διαδικασιών για να τους βοηθήσει. Πρόταση λοιπόν, κοιτάξτε την. Άρθρο 6-7, μορατόριουμ, καθώς και επιπτώσεις του μορατόριουμ, της αναβολής ή της αναστολής. Προβλέπει η πρόταση οδηγίας ένα μορατόριο με συγκεκριμένες επιπτώσεις. Εγώ θεωρώ θετικό ότι υπάρχει το μορατόριουμ αυτό, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν και κάποιο περιθώριο να αναπνεύσουν, δηλαδή να μπορέσουν και να σκεφτούν έχει νόημα να κάνω το α ή το β, τι μπορώ να κάνω, να διεξαχθούν συζητήσεις. Αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα. Νομίζω πάντως ότι σε αυτό το στάδιο της προδικασίας, της προδικασίας ας πούμε, αυτό θα πρέπει να επιταχυνθεί, να περιοριστεί η διάρκεια του μορατόριου σε ένα δίμηνο, με την δυνατότητα ωστόσο να παραταθεί έως ένα ανώτατο όριο εξαμήνου. Εφόσον όμως υπάρχει αφαιρεγγιότητα, θεωρώ ότι προς το συμφέρον των πιστωτών πρέπει να γίνει αίτηση για αναγνώριση αφαιρεγκαιότητα. Έχω το άρθρο 7 μετά για τις επιπτώσεις του μορατόριου. που θα πρέπει να ε, μπορεί να καταγγείλει άλλες συμβάσεις εκτός από τις ουσιώδεις ή τις θεμελιώδεις. Δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινά το μορατόριο διακόπτεται κάθε δραστηριότητα, αλλά πρέπει να τηρούνται οι δεσμεύσει που έχουν αληφθεί έως τώρα, έως τη στιγμή εκείνη. Θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση εκεί. Θα πρέπει αυτή η de facto υποχρέωση του προμηθευτού να παρέχει τα ε, αναγκαία να υπάρξει μονάχα για τις ουσιώδεις συμβάσεις. Αυτά το 9 έως 11 αναφέρονται στην αποδοχή και αναγνώριση των σχεδίων αναδιαρθρώσεως. Θα πρέπει οι πιστωτές να έχουν δυνατότητα να ψηφίζουν τα σχέδια αυτά αναδιαρθρώσεως. Είμαι πεπισμένη ότι χρειάζεται τουλάχιστον η πλειοψηφία των πιστωτών να συμφωνήσουν δηλαδή υπέρ του σχεδίου αναδιάθρωσης, διότι εν τέλει κανείς δεν εξυπηρετείται ε, να λαμβάνονται αποφάσεις πίσω από τις πλάτες των ενδιαφερομένων. Και για τον λόγο αυτό έχω και το μειώσει κάπως, έχω περιορίσει κάπως το περιεχόμενο του άρθρου 11, διότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης μπορούν αποτελεσματικά μόνο όταν τα στηρίζει η πλειοψηφία των ε, πιστωτών. Βλέπετε ότι προβλέπω κάποιες τροποποίησεις στο σχέδιο της Επιτροπής που ενισχύουν την θέση των πιστωτών. Εξετάστε τα. Τελευταίο, άρθρα 19-23. Απαλλαγή από τα χρέη. Θεωρώ ότι για την πλήρη απαλλαγή από το χρέος του επιχειρηματία. Αυτή έχει κάποιο νόημα και αποτελεί τη δυνατότητα για μια νέα ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία μετά από την αποτυχία. Θα πρέπει να είναι στόχος μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή αποτύχει μια πρώτη επιχείρηση, όπως είπα, να μην κουβαλάει ο άνθρωπος αυτός, ο επιχειρηματίας, το στίγμα σε όλη τη ζωή. Αυτό είναι σημαντικό. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, η αποτυχία σε μια πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται κάτι τι το αυτονόητο. Από αυτά μαθαίνουν οι άνθρωποι. Ενώ εδώ ε, είναι βαρύτατο το στίγμα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι εδώ πρέπει να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί μια ε, νοοτροπία η οποία ε, θα σημαίνει, θα δείχνει ότι η αποτυχία ενδεχομένω αποτελεί και ένα πρώτο δίδαγμα. Υποστηρίζω τη δυνατότητα της χώρας μέλους να συνδέσει την απαλλαγή από τα χρέη με κάποιες πληρωμές που θα πρέπει να κάνει ο υπεύθυνο, πάντοτε όμως υπό το κριτήριο του έντιμου επιχειρηματία. Δηλαδή, ο φιλέτης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει καλή πίστη. Άρα, η απαλλαγή από τα χρέη θα συνδέεται με ορισμένες πληρωμές και για την πρώτη απαλλαγή νομίζω ότι ένα περιθώριο τριών ετών είναι κατάλληλο μια ε, διάρκεια δηλαδή τριών ετών και μετά να χορηγείται απαλλαγή. Εάν αποδειχθεί ότι έγινε καταχρηστική πρόσβαση στην απαλλαγή από τα χρέη, τότε θα πρέπει για την επόμενη φορά να ισχύσουν πολύ αυστηρότερες διατάξεις. Ολοκλήρωσα εδώ την παρουσίαση του κειμένου μου. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση και εδώ στην Επιτροπή αλλά και στο ακόλουθο χρονικό διάστημα. Όπως είπα είναι περίπλοκο το θέμα προσπάθησα να εξισορροπήσω με τον τρόπο που μου φάνηκε πιο σωστός τα διάφορα, καμιά φορά και αντιτιθέμενα συμφέροντα και θέτω πάντως ε, το πόνημά μου υπό την κρίση σας. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Νίμπλερ για την πληρέστατη ε, ανάπτυξη του θέματος, πολύ ενδιαφέρουσα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοφεράτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Εγώ πιστεύω πως όταν βρίσκεται κάποιος σε μία κρίση βαθιά όπως αυτή που έπληξε την Ευρώπη και συνεχίζεται ακόμη σε ορισμένες χώρες, είναι χρήσιμο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ορίσουν ποια είναι τα κατάλληλα μέσα παρέμβασης στην κρίση αυτή με στόχο να δοθεί όθηση στην παραγωγική διαδικασία. Δεν πρέπει να είμαστε παθητικοί, αλλά πρέπει να βρούμε τις ε, αιτίε και να εντοπίσουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να περασπίσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης που είναι σε δυσκολία, αλλά κυρίως πριν από την τελευταία εγγύηση, δηλαδή πριν από την διαδικασία φερεγγιότητας να έχουμε όλες τις κατάλληλες διαδικασίες για την αναδιάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας. Το δεύτερο στοιχείο γενικού χαρακτήρα που θέλω να υπογραμμίσω είναι το εξής. Για να μπορούμε να το κάνουμε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία αναδιάρθρωσης και να έχει και θετική έκβαση, πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει μέγιστη διαφάνεια και μέγιστη μπλοκή από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διαφάνεια για να αποφύγουμε να υπάρχει κακή διαχείριση που στη συνέχεια θα ποινικοποιήσει τους πιο αδύναμους, αλλά και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών, γιατί η δική τους ε, άποψη μετράει, είναι πολύ σημαντική, γιατί τα, οι συνέπειες θα βαρύνουν τους ιδίους. Είναι θετική, θετική η σκοπή της Κομισιόν, όπως είπα, και μάλιστα είχαμε και κάποια σχόλια από την εισηγήτρια. Εμείς θα παρουσιάσουμε τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί πιστεύω ότι πολλές ε, πτυχές από την πρόταση της Κομισιόν μπορούν να βελτιωθούν. Έλεγα λοιπόν ότι ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος για να γίνει όμως θα πρέπει να εμπλακούν όλοι και μάλιστα προληπτικά. Όχι όταν θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία φερεγγιότητας, αλλά εκ των προτέρων. Όταν θα διαπιστωθούν οι συνθήκες. Θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως και για τους εργαζομένους. Προληπτική εμπλοκή λοιπόν, προληπτική συμμετοχή. Ξέρω ότι ασχολήθηκε με αυτό το θέμα η συγγήτρια, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το σημείο και να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Κατόπιν, οι πιστωτέ δεν είναι όλοι ίσοι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Πιστεύω, όπως λέει και η Κομισιόν που θέλει να διακρίνει μεταξύ των κατηγοριών των πιστωτών, πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτών που δεν καλύπτονται από εγγύηση και των υπολείπων. Αλλά στη συνέχεια πρέπει να δούμε και τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση των εργαζομένων. Σε αυτή την κατηγορία υποχρεωτικά πρέπει να δώσουμε δικαιώματα, γιατί ε, αντικειμενικά είναι οι πιο αδύναμοι. Θα πρέπει να προστατευτούν από την ομοθεσία. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν και μια αποζημίωση. Δεν θα πρέπει να φυγεί ο μισθός τους κατά την περίοδο αναστολής. Διαφορετικά Μπορεί να έχουμε εδώ πέρα μια θετική πρόθεση, αλλά θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Στη συνέχεια υπάρχει μια συγκεκριμένη πτυχή που αφορά ένα από τα χαρακτηριστικά της οικονομικής ε, κρίσης ε, που ακόμα πλήττει πολλές χώρες όπως σας είπα και αφορά το ατομικό χρέος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταστήσουμε υποχρεωτικό για τα ατομικά χρέη να προβλέπονται μέσα αναδιάρθρωσης. Όχι, όπως ε, λέει η Κομισιόν, ε, να το ορίσουν τα κράτη-μέλη. Στην οδηγία θα πρέπει να ορίζεται αυτή η υποχρέωση να προστατεύουμε τα ατομικά χρέη. Και τέλος, όπως σας είπα, αξιολογούμε το έργο της εισηγήτριας. Όμως υπάρχουν δύο πράγματα στα οποία είμαστε αντίθετοι εμείς. Το πρώτο είναι δεν βρίσκουμε ούτε χρήσιμο ούτε δίκαιο να ξεκινήσουμε την επίσημη διαδικασία αφαιρεγγιότητας κατόπιν ετήματος των πιστωτών κατά τη διάρκεια της αναστολής οι πιστωτέ πάντοτε θα είχαν συμφέρον να το κάνουν, γιατί θα υποφελούνταν, όμως όλοι οι υπόλοιποι θα ποινικοποιούνταν. Και το δεύτερο σημείο αντίθεσης αφορά τη μέγιστη περίοδο αναστολής. Η πρόταση της Κομισιόν μου φαινόταν λογική. Τέσσερις μήνες που το πολύ θα μπορούσαν ε, να φτάσουν στους 12. Άκουσα τα επιχειρήματά σας και κατάλαβα γιατί θέλετε μείωση της περίοδου αυτής. Όμως να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την διαδικασία και ιδίω τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι δύο μήνες που προτείνεται είναι πάρα πολύ λίγοι. Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να διατηρήσουμε την αναφορά στην περίοδο που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερις μήνες δηλαδή, με μέγιστη παράταση μέχρι τους 12 μήνες. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, θα τις παρουσιάσουμε, θα τις συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ, όπως και να έχει, για την ε, προσέγγισή σας για ένα θέμα που αναγνωρίσετε κι εσείς είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έχει τεχνικές στοιχές ιδιαίτερα πολύπλοκες και ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ λεπτό θέμα γιατί αφορά τις ε, επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ένα δύσκολο στάδιο και τους πιο αδύναμους ανθρώπους. Όμως ε, θα τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Thank you. Η Πρόεδρος, κυρία Ντελβό, ευχαριστώ Σέζιο, η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένη ότι είναι σε καλά χέρια το θέμα. Είμαι Βεβαίω ότι η κυρία Νίμπλερ έχει πραγματικά εμβαθύνει στο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και εύκαμπτο πλαίσιο για την αναδιάρθρωση. Για μια ενιαία αγορά η οποία είναι όλο και πιο ολοκληρωμένη. Είναι σημαντικό επίσης για να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στους έντιμου επιχειρηματίες να αποφευθεί ώστε ορισμένοι ενδεχομένω να αισθανθούν τον πειρασμό να πάνε σε, κατευθυνθούν πιο πολύ σε, μια, σε κάποιους γκρίζους ή και μαύρους τομείς της οικονομίας. Αυτά θα ήθελα να πω για την ώρα. Θα εξετάσουμε σε συνεργασία με την κυρία Νίμπερ κάποιες λεπτομέρειες, αλλά αρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Χάουταλα. Ο κύριος Μαρίνιου Επίντου. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πρώτος ο κύριος Ράντεφ. Ε, να με, να με συγχωρείτε κύριε Μαρίνιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Νίμπλερ για το σχέδιο εκθέσεως για την ε, έκθεσή της για την προβλητική αναδιάρθρωση και τη δεύτερη ευκαιρία. Ως δικηγόρος και σύνδικος στοχεύσεων το να δοθεί Λέγω ότι το να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις είναι σημαντικό βήμα προς τα μπρος, το οποίο θα ενισχύσει την οικονομική ζωή, τις ευκαιρίες των επιχειρηματιών, θα μπορέσουν να, να ελαφρυνθεί το χρέος πολλών φυσικών προσώπων, διότι η υπερχρέωση πολλών φυσικών προσώπων αποτελεί σημαντικό πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα. 11,4% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν τα προστοζήν κάθε μέρα. Η ρύθμιση αυτή θα επιτρέψει επίσης να μην χάσουν τα λεφτά τους οι πιστωτές όταν ρευστοποιηθεί η επιχείρηση που έχει πτωχεύσει. Και να μην βαρύνει έτσι και τον ισολογισμό των πιστοτικών ιδρυμάτων θεωρώ ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των πιστωτών και των οφειλετών. Οι πιστωτές, ας μην το λησμονούμε, μπορεί να είναι και οι ίδιοι ευάλωτες μικρές επιχειρήσεις. Το δικαστήριο είναι βεβαίως ο καλύτερος εγγυητής της ισορροπίας αυτής. Γι' αυτό και νομίζω ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να μπορέσουν οι ίδιες να ρυθμίσουν το ρόλο του δικαστηρίου στην ε, διαδικασία της αναδιάρθρωσης. Άλλο σημαντικό θέμα είναι του ορισμού επαγγελματία, εμπειρογνώμονα δηλαδή, αναδιαρθρώσεων. Εδώ θα πρέπει να φανούμε ευέλικτοι, να λάβουμε υπόψη τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων ενόμων τάξεων και να δράσουμε κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης και του οφειλέτου και των οικονομικών πόρων που ενδεχομένως να διαθέτει και του είδους επιχειρήσεως και ελπίζω θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή ισορροπία των στόχων μας που να ικανοποιεί και τους οφειλέτες και τους πιστωτές. Ευχαριστώ κύριε Ράντεφ. Τώρα ο κύριος Μαρίνιο Επίντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο πολύ σύντομα σχόλια για το θέμα αυτό. Καταρχήν, Φυσικά να δηλώσω την εμπιστοσύνη μου στην εισηγήτρια και στην εξαιρετική δουλειά της. Δεύτερον, θέλω να πω ότι συμφωνώ και προσυπογράφω την πρόταση του συναδέλφου Κοφεράτη για το να αναφέρουμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τους μισθωτούς σε μια διαδικασία φεραγγιότητας. Δηλαδή πρέπει πάντοτε να προστατεύουμε τον πλέον αδύνατο σε αυτή τη διαδικασία και ποιο είναι ο πλέον αδύνατος εδώ, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται μπροστά στην προοπτική της ανεργίας. Όμως υπάρχει και ε, ένα άλλο θέμα για το οποίο θέλω να κρούσω τον κοδόρα του κινδύνου, ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορεί να πτωχεύσουν, ε, δηλαδή λόγω ε, του θέματος που συζητάμε. Παραδείγματο χάρη, ε, εγώ ε, ως δικηγόρος συμμετείχα σε πάρα πολλές επιτοθετικές διαδικασίες και ουσιαστικά πολλές επιχειρήσεις που είχαν χρεοκοπήσει δεν μπορούσαν να πληρώσουν άλλες επιχειρήσεις φυσικά οι πιστωτές ε, είναι αυτοί που θέτουν τους κανόνες και συνήθως είναι οι μεγάλες τράπεζες. Είναι το χρέος στις τράπεζες που ουσιαστικά ε, θέτει τη δαμάκλειο σπάθη πάνω από την επιχείρηση που έχει χρεοκοπήσει. Πολλές ε, φορές όμως ε, τα συμφέροντα αυτών είναι αντίθετα από τα συμφέροντα ανθρώπων που εργάζονται στην πραγματική οικονομία. Είναι αντίθετα στα συμφέροντα της οικονομίας που συνεισφέρει στην ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, και κερδοσκοπικά στοιχεία στο χρηματοοικονομικό κεφάλαιο που δεν συνάδουν με την οικονομική ανάπτυξη. Εγώ λοιπόν ήθελα να σας προειδοποιήσω για το θέμα αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις που μπορεί και αυτές ε, να χρεοκοπήσουν. Δηλαδή μια χρεοκοπία μιας άλλης επιχείρησης να επιφέρει και τη δική του χρεοκοπία. Ευχαριστώ, κύριος Λεμπρετών. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Νίμπλερ που ασχολείται με αυτό το σημαντικό φάκελο. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, χρεοκοπίες των επιχειρήσεων που ήταν ε, και πολύ άρθιμες τελευταία. Είναι αξιέπαινος ο στόχος, ε, όμως Έχω κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, θέλουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των πιστωτών αλλά και του προσωπικού. Μεταξύ των ε, τροπολογιών ε, είχαμε πολλές που υπερασπίζουν ε, τον πλέον αδύναμο κρίκο, δηλαδή τα συμφέροντα των πιστωτών. Πιστεύω ότι αυτή η ιδέα της δεύτερης ευκαιρίας είναι ενδιαφέρουσα για να επιτρέψουμε σε κάθε επιχειρηματία ε, μετά από μια πρώτη αποτυχία ε, να μπορέσει ε, να προσπαθήσει να τα ξανακαταφέρει. Και έχω μία σειρά ερωτηματών. Κάνετε μία διάκριση μεταξύ του έντυπου επιχειρηματία και του άλλου προσπαθεί να καταχραστεί τη διαδικασία της αφαιρεγγιότητας. Δεν θα είναι εύκολο να κάνετε αυτή τη διάκριση θα πρέπει <laughs> να εργαστείτε από αυτού. Είπατε μάλιστα κυρία Νίμπλερ ότι θέλετε συγκεκριμένους κανόνες για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και εδώ νομίζω ότι προς στιγμή ε, δεν είναι όριμη η πρόταση και εδώ θα πρέπει να εργαστούμε. Για την διάρκεια της αναστολής ε, προτείνεται από τους τέσσερις μήνες να πάμε στους δύο μήνες εδώ. Θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να έχουμε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για διαδικασίες που χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Δύο παρατηρήσεις για να κλείσω. Καταρχήν να πω ότι δεν κατάλαβα ένα μέρος της παρέμβασης του κυρίου Κοφεράτη. Φαίνεται ότι προτείνατε να διευρυνθεί το κείμενο για να βάλετε και το θέμα των προσωπικών των προσωπικού χρέους αν πρόκειται για κάτι τέτοιο, εγώ δεν είμαι υπέρ, ίσω να μην κατάλαβα. Ή κατάλαβα, μπορεί και να κατάλαβα. Και σε ό,τι αφορά την ε, απαραίτητη ευελιξία που ανέφερε ο κύριος Ράντεφ, δεν θα ήθελα το κείμενο να καταλήξει σε μεγάλη ομογενοποίηση σε επίπεδο κρατών μελών. Θα πρέπει να αφήσουμε και μια ευελιξία σε κάθε κράτος μέλος. Σας παρακαλώ, σκεφτείτε παρακαλώ και την εθνική κυριαρχία γιατί η ομογενοποίηση δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνει πολύ μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η δεύτερη ευκαιρία είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική έννοια για τις επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους γεωργούς. Είναι εξαιρετική η δουλειά της κυρίας Νίμπλερ και νομίζω ότι είναι πραγματικά θεμελιώδες για την οικονομία μας το ΚΕΜΠΕΡ, α πούμε, 60.000 κάτοικοι, 700 πτωχεύσεις κατ' έτος, ε, προς, ξέρω λοιπόν γιατί μιλάμε και θα ήθελα να συμφωνήσουμε τι εννοείται ε, φερεγγιότητα, γιατί δεν μιλάω για μία ε, επιχείρηση ε, παροχής υπηρεσιών. Σκέφτομαι κυρίως τους γεωργούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάσουν σπίτια, μεγάλες επιχειρήσεις επίσης, μία επιχείρηση η οποία εγκαθίσταται κάπου, έχει, είναι από την αρχή αφαιρέγγια γιατί αγοράζει τον εξοπλισμό της, αγοράζει τις ε, μηχανές αν δεν έχει απόδοση η επιχείρηση αυτή, αν δεν έχει κέρδο, σε 5-6 χρόνια θα αποδοχεύσει. Η διαφορά λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ε, του, της πίστοσης και του leasing, της εκμίσθωσης. Το leasing είναι μια, ε, ένα κίνητο ε, το οποίο σήμαινε ότι όλο και περισσότεροι ε, ιδιοκτήτες υπήρχαν για ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Οι τράπεζες όμως τα κατάφεραν κατά τέτοιο τρόπο ε, είναι η, μηχανή η οποία πληρώθηκε κατά 89% ανήκει ακόμη στην ε, τράπεζα και δεν μπορούμε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στο γεωργικό που το τρακτέρ του έχει χαλάσει οι τράπεζες επειδή θεωρητικά παραμένουν ιδιοκτήτριες ξαναπαίρνουν ε, πίσω όλες τις ε, όλα τα, τα μέσα της παραγωγής. Όχι μόνο οι τράπεζες αυτές παραμένουν ιδιοκτήτριες ε, του αγαθού το οποίο έχει αγοραστεί, αλλά ε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος που το έχει αγοράσει, ο ίδιος πρέπει να δεσμευτεί, να πληρώσει την τιμή, ε, ενώ ήδη δεν έχει τα μέσα και δεν υπάρχει περίπτωση να αποζημιωθεί και φυσικά οι εργαζόμενοι του βρίσκονται όλοι στην ανεργία. Για μένα το βασικό είναι αυτό. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Αυτό το σύστημα του leasing που όλο και περισσότερο αντικαθιστά το δάνειο το απλό, ε, μερικές φορές με εγγύηση, ε, με απόσβεση, αλλά που δεν δίνει τη δυνατότητα ε, στην τράπεζα, που δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα να ζητήσει πίσω αυτό το οποίο είναι ιδιοκτήτρια. Ε, πρέπει δηλαδή να μπορούμε να πούμε ότι οι μικρές αυτές ρήτες που λένε ότι αυτός που έχει αγοράσει τη μηχανή θα είναι ιδιοκτήτης μόνο αυτή τη στιγμή ε, θα έχει καταβάλει τα 2.000 ευρώ που παραμένουν μετά την τελευταία, το τελευταίο νίκη. Ε, τι να σας πω, ε, τελικά ε, καταλήγουμε σε επιχειρήσεις που δεν υπάρχει καμία απολύτως μηχανή πια και δεν υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία να τους καλύψει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να στραφώ τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της. Ε, εμείς ε, εκτιμούμε όλος ιδιαίτερο την υποστήριξή σας ε, για πολλές από τις προτάσεις μας και ειδικότερα την δεύτερη ευκαιρία για τους έντιμους επιχειρηματίες. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό είναι ένα τεράστιο τμήμα της πρότασής μας. Ε, θα υπάρχουν βεβαίως ε, δυσκολίες, ε, διάκριση μεταξύ του έντιμου και του ανέντιμου επιχειρηματία, αλλά υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θέσουν κάθε είδους περιορισμούς για να αποφύγουν εκείνοι που είναι ανέντιμοι και που είναι μια μικρή μειοψηφία κατά τη γνώμη μου, να μην μπορούν να καταχρώνται του συστήματος. Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις που έγιναν για το κεφάλαιο αναδιάρθρωσης ε, που ε, θα βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό το κείμενο. Επιτρέψτε μου επίσης ε, να σχολιάσω μερικές μόνο προτάσεις για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε κάπως τη δική μας προσέγγιση. Καταρχάς προτείνεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας κοινό ορισμός για την πιθανότητα αφηρεγγιότητας. Δεν το λέτε μόνο εσείς, το έχουμε ακούσει και από άλλους, από τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παράδειγμα. Ε, θα συμφωνούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά αυτό που είναι πολύ δύσκολο είναι να υπάρχει ένας ορισμός για την πιθανότητα αφαιρεγγιότητας, απουσία ορισμού περιφερεγγιότητας. Ε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε την αφαιρεγγιότητα ναι, ομοιόμορφα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν ε, δύσκολο να ε, εναρμονίσουμε και το τι θα πει πιθανότητα αφαιρεγγιότητας. Η απειλή για τη ρευστότητα και η σχετική τροπολογία Ενδεχομένως σε κάποια κράτη-μέλη αυτό μπορεί να σημαίνει αφαιρεγκαιότητα. Σε μερικά κράτη-μέλη αυτό ε, δρομολογεί ε, τη διαδικασία εκαθάρισης λόγω αφαιρεγγιότητας. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, θα είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε επί ενός κοινού ορισμού μεταξύ των κρατών μελών, τουλάχιστον αυτό τι ήταν ε, η λογική μας όταν αποφασίσαμε να μην υπάρχει ε, πρόταση για έναν τέτοιο κοινό ορισμό. Για τη διάρκεια, ε, τη μεγάλη διάρκεια για τη μεγάλη διάρκεια αναστολή. Ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός που θα είναι κοινό ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θα είναι δύο μήνε, τρει μήνε, τέσσερις μήνε. Αυτό είναι συζητήσιμο. Κατά τη γνώμη μας, ε, βάσει αποδεκτικών στοιχείων από τα κράτη-μέλη ε, κατά τις, προ, κατά τις πρόσφατες, μετά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, τέσσερις μήνες ε, είναι η καλύτερη λύση. Βέβαια τα κράτη-μέλη μπορεί να αποφασίσουν ε, ένα συντομότερο χρονικό διάστημα, αλλά οι δύο μήνες ε, νομίζω μόνο σε ένα ή δύο κράτη-μέλη υπάρχουν. Οπότε... Από την πείρα μου θα έλεγα, τέσσερις μήνες αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών. Ένα ακόμη τεχνικό ζήτημα ε, που αφορά τους περιορισμούς ε, για τη χώρα στην οποία έχει εγκατασταθεί ο επιχειρηματίας ε, είναι ένα πρόβλημα τους τελευταίους μήνες. Το πρόβλημα είναι η αλλαγή ε, του αναθεωρημένου κανονισμού περιαφερειγιότητας ε, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις για αυτή την περίπτωση όταν μια ε, εταιρεία μετεγκαθίσταται από τη μία χώρα στην άλλη. Εδώ βλέπουμε ένα πρόβλημα σύγκρουσης με τον κανονισμό αυτό. Άρχισε να ισχύει μάλιστα πριν από μερικούς μήνες και θα είναι δύσκολο και πρόημο να αλλάξουμε την προσέγγιση για τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν την έγκριση του σχεδίου από τους πιστωτέ, ε, όπου αναφέρεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει διπλή πλειοψηφία δηλαδή και για την αξία ε, αλλά ε, και στον αριθμό των πιστωτών αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα καθιστούσε πιο δύσκολη την έγκριση του σχεδίου, αλλά δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη με καλά συστήματα αναρδιάρθρωσης που δεν έχουν αυτή τη διπλή ε, πλειοψηφία. Οπότε θα προτείναμε λίγη ευελιξία για αυτά τα κρατη που να τους επιτρέπει να κρατήσουν ε, το σύστημα απλής πλειοψηφίας ε, κατά την έγκριση αυτών των ε, σχεδίων διάρθρωσης Όσον αφορά το cross-class crumb-down». Ε, συμφωνώ ότι για τους πιστωτές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν όμως το πρόγραμμα, το σχέδιο αναδιάρθρωσης υποστηρίζεται από μία τάξη πιστωτών, θα πρέπει αυτό να είναι επαρκές ε, για να μπορεί το δικαστήριο να ε, το εγκρίνει και με κάποιες άλλες διατάξεις ε, ισχύει αυτό, κάποιες ευέλικτες διατάξεις που υπάρχουν ε, σε κράτη-μέλη με ψηλές επιδόσεις, που έχουν πολύ καλά ε, σχέδια αναδιάρθρωσης. Θα, αν ένας πιστωτός είναι καλύτερο στο πλαίσιο μιας ενός μιας αναδιάρθρωσης, ε, τότε αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης θεωρείται καλό και πρέπει να μπορούμε να διατηρήσουμε αυτή την ευελιξία. Το άρθρο 11 την επιτρέπει. Λέμε ότι το πρώτο άρθρο, στο άρθρο 1 λέει ότι ε, υπάρχει αυτή η τάξη που αποφασίζει και μετά λέμε στο δεύτερη, στη δεύτερη παράγραφο ενδεχομένως και περισσότερες ε, κατηγορίες. Ε, μπορούν να υπάρχουν και ε, θα θέλαμε να μπορούμε να διατηρήσουμε όλες αυτές τις λύσεις ε, που λειτουργούν καλά. Ένα ακόμη ερώτημα που ετέθη από πολλούς σήμερα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας εξηγήσω το εξής. Εξετάζοντας το τι υπάρχει στα κράτη-μέλη, εμείς πιστεύουμε ότι μια ειδική διαδικασία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να μην είναι πολύ χρήσιμη. Δεν υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν ειδικέ διαδικασίες ε, μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεπώς δεν έχουμε κάνει σχετική πρόταση. Αυτό που προτείναμε όμως είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι ευέλικτη και θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες και και των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωστόσο δεν διαφωνούμε με το να εφαρμόζουν την οδηγία τα κράτη-μέλη και ε, μέσω μιας διαδικασίας ταχείας και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί κατά την εφαρμογή της ε, οδηγίας. Για τους ε, εργαζομένους έχουμε προβλέψει μία σειρά μέτρων που έχουν ε, βελτιώσει ή θα βελτιώσουν τα δικαιώματά τους, ότι η αναστολή δηλαδή δεν θα επηρεάσει τους τις αξιώσεις ε, των ε, εργαζομένων. Επίσης, έχουμε προβλέψει στην πρότασή μας ότι όταν ένα σχέδιο αναδριάρθρωσης επηρεάζει τους, ε, τις μελλοντικέ αξιώσεις των μελλοντικών εργαζομένων, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν και θα έπρεπε να αποτελούν και μια ξεχωριστή κατηγορία, να μην να μην ε, υπερψηφιστεί κάτι από τους υπόλοιπους πιστωτές ε, και δεν ληφθούν υπόψη. Ε, αυτά λοιπόν περί προστασίας εργαζομένων. Για τις τράπεζες, αυτό που έχουμε κάνει ε, στην πρόταση αυτή είναι να τους συμπεριλάβουμε στη διαδικασία αναρδιάρθρωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπου οι ασφαλείς πιστωτές δεν συμμετέχουν στην αναδιάρθρωση και ε, συνεπώς ε, ε, η θέση τους δεν μπορεί να αλλάξει κατά κανέναν τρόπο. Εμείς θέλουμε αυτοί οι πιστωτές να μπορούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση σε όλα τα κράτη-μέλη και μπορούν να δεσμεύονται από ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Θα σταματήσω εδώ. Υπάρχουν ε, και άλλα ε, σχόλια ε, ενδεχομένως, αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο, πολύ χρόνο, για να συζητήσουμε τις διάφορες τροπολογίες. Αγαπητή Αγγέλικα, θέλετε να προσθέσετε κάτι ή να πείτε, να, δηλαδή να λάβετε τη τελευταία το λόγο. Ναι, δεν θέλω να αφήσω το τελευταίο λόγο στην Επιτροπή, ασφαλώς όχι. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους, καθώς και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να ευχαριστήσω λοιπόν όλα τα πρόσωπα αυτά για τις παρατηρήσεις τους. Και χαίρομαι πολύ που αρχίζει η συζήτηση τώρα και όταν θα φτάσουμε στις επιμέρους τροπολογίες. Έρχομαι κάπως αθαίρετα σε ορισμένα ζητήματα που μου φάνηκαν πιο ενδιαφέροντα. Αφενός, πόσο εύκαμπτη πρέπει να είναι η οδηγία η Κομισιόν δικαίως τονίζει ότι δεν υπάρχει κοινό ορισμός για την έννοια ε, αφαιρεγγιότητα σε όλες τις χώρες μέλη. Οφείλουμε πάντοτε σε οποιοδήποτε νομοθέτημα ε, να σκεφτόμαστε ε, θα αφήσουμε τις χώρες μέλη να έχουν την ευχέρεια, τη διακριτική ευχέρεια ή θα το ρυθμίσουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μας απασχολήσει και εδώ. Για το επόμενο θέμα, ιδιωτικά χρέη. Κύριε Κοφεράτη, εσεί το θίξατε το θέμα αυτό και εγώ το έχω περιλάβει στο σχέδιο εκθέσεώ μου ότι οι χώρε μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν θα περιλάβουν και τι αφαιρεγκαιότητα και πτωχεύσει προσώπων, τι ατομικέ, τι ιδιωτικέ δηλαδή. Αυτό θα δούμε αν θα γίνει υποχρεωτικό ή όχι. ένα θέμα λοιπόν για το ζήτημα της αναστολής του μορατόριου και της διαρκείας του τα λέω κάπως σύντομα, δεν μιλούμε ε, να γίνει μια πλήρης εξυγίανση μια επιχειρήση γιατί κάτι τέτοιο χρειάζεται χρόνια. Ε, ρωτούμε εδώ πόσο καιρό θα πρέπει να ισχύει το μορατόριο, δηλαδή οι πιστωτέ θα πρέπει να χορηγούν τα υπεσχημένα, προμηθευτέ κλπ, ενώ δεν ε, παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Αυτό ακούσαμε την άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τετράμινο ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια. Για τις μικροεπιχειρήσεις παραμένω ανοιχτή σε προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε μόλις γιατί έχει αφήσει τις ΜΜΕ εκτός πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό θα το λύσουν υποτίθεται οι χώρες μέλη. Η ερώτηση δική μου είναι να το περιλάβουμε, τότε όμως πρέπει να ξαναδούμε ολόκληρο το κείμενο της οδηγίας. Τι θα ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι όχι. Ή θα κάνουμε αυτό λοιπόν, με πλήρη επανεξέταση της ε, οδηγίας ή θα τα αφήσουμε στις χώρες μέλη για τις μικρές, πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις ή και ε, μικροεπιχειρήσεις. Για τον έντιμο επιχειρηματία, πάλι εκεί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια ε, να βρω κάποια λύση. Ε, θεώρησα ότι ένα κριτήριο μπορεί να είναι η ε, νόμιμη τήρηση, ορθή δηλαδή τήρηση σύμφωνα με τον νόμο των λογιστικών βιβλίων. Αυτός λοιπόν τότε είναι έντιμο επιχειρηματία. Αλλά είμαι ανοιχτή και εδώ, αν υπάρχουν και άλλα κριτήρια, αν μπορούμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο, τόσο το καλύτερο. Η περίπτωση που θίγει η κυρία Μπεζερόν. Αγαπητή κυρία Μπεζερόν, το έχετε ε, επισημάνει αυτό και άλλη φορά στην πρώτη μας συζήτηση, ομολογώ ότι δεν ξέρω πώς μπορούμε να το λύσουμε. Όταν δηλαδή τα μηχανήματα, τα μέσα της παραγωγής ε, διατίθενται με την επιφύλαξη της κυριότητας, ε, τότε βεβαίως την κυριότητα την κρατάει ο προμηθευτής του μηχανήματος μέχρι την πλήρη εξοφλησή του. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή. Έκανα μεγάλη προσπάθεια να βρω κάποιες λύσεις το πρόβλημα που έχετε εξηγήσει το έχω καταλάβει καλά. Ομολογώ ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να περιληφθεί στην οδηγία. Πολύ ευχαρίστω όμως θα ακούσω προτάσεις από εσά. Το τελευταίο, έρχομαι στον κύριο Ράντεφ, για, μας, όντως, για μένα όμως το σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ισορροπία. Να εξορροπηθούν τα ε, συμφέροντα των πιστωτών και των οφειλετών και βεβαίω εδώ εντάσσονται και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Όπως είπε και ο κύριος Ντεπίντο, που πρέπει να τα έχουμε διαρκώς υπόψη μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γράψει πολλά σχετικά. Εγώ έχω περιλάβει δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πληροφόρησης των εργαζόμενων. Να μου πείτε αν σας αρκεί αυτό ή όχι. Δεν μιλούμε ακόμη για την αφαιρεγγιότητα. Είναι σαφές ότι σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας ε, πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μιλούμε για την προκαταρκτική φάση της διαδικασίας όπου ε, ακόμα ισχύει και ένας εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών αυτών. Θα δούμε. Ευχαριστώ όλες και όλους για τις πρώτες αυτές τις παρατηρήσεις, οι οποίες ε, μου δίνουν μια πρώτη εντύπωση σχετικά με την πορεία που θα θέλετε να λάβει η συζήτηση και αναμένω βεβαίως με ενδιαφέρον και τις υπόλοιπες ανταλλαγές απόψεων. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, κυρία Πρόεδρε, βρίσκομαι στα χέρια σας. Μπορώ να προσθέσω μόνο, λέει η πρόεδρος κυρία Ντελβό, είναι ότι η προθεσμία ε, τροπολογιών η 7η Νοεμβρίου, η Ενδεκάτου στις 12 το μεσημέρι. Και μετά γίνεται κάπως πιο περίπλοκο το θέμα, δεν θα σας πω τίποτε άλλο. Νομίζω λοιπόν ότι καταλήξαμε σήμερα, τελειώσαμε δηλαδή, εξαντλήσαμε την ημερησία διαταξή μας. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής θα είναι στις 20 Νοεμβρίου, Δευτέρα και Τρίτη 21. Και μετά έχουμε και μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις, ε, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο. Πάντοτε σημαντική προσέλευση ε, στο Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ και καλό σας βράδυ.